So welcome everyone. We will... Καλώς ορίσατε. Θα αρχίσουμε πάνω κάτω στην ώρα μας για αλλαγή σήμερα. Ε, σημείο πρώτο στην ημερήσια διάταξη έγκριση αυτής. Δεν βλέπω κανείς να διαφωνεί. Είμαστε εντάξει, ωραία. Έγκριση των πρακτικών είναι το δεύτερο σημείο των συνεδριάσεων ε, των εξή ημερομιών. 20 ε, ε, Φεβρουαρίου 2014, 24 Φεβρουαρίου 2014 και 3 Μαρτίου 2014. Εξ όσων βλέπω δεν διαφωνεί κανείς, εγκρίνονται και τα πρακτικά και πάμε αμέσως τα βασικά θέματα σήμερα σε διάταξη σήμερα που είναι η πιθανή υιοθέτηση του ευρώ τη Λιθουανία, ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό και το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Λιθουανίας. Θα ήθελα να καλωσορίσω ε, τον Υπουργό και τον διοικητή ε, στα πλαίσια αυτή τη συζήτηση για την πιθανή οθέτηση, όπως είπαμε, του ευρώ από τη Λιθουανία. Από ό,τι ξέρετε, είναι η επόμενη ε, χώρα που προαλήφεται να μπει στο ευρώ 1η Πρώτου 2015. Έχουμε τη χαρά σου και την τιμή σήμερα λοιπόν να φιλοξενούμε τον Υπουργό Οικονομικών ε, της Λιθουανίας και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Βέβαια ε, την ε, επίσημη απόφαση θα τη λάβει το επόμενο κοινοβούλιο και η Επιτροπή Οικονομικών του, αλλά εμείς έχουμε κάνει ουσιαστικότατα την προετοιμασία. Με άτυπη ε, κοινοβουλευτική δουλειά και εισηγητή τον κύριο Βέρνερ Λάγκε. Στις 7 Απριλίου θα παρουσιάσει την έκθεσή του, άτυπη επαναλαμβάνω, που δεν θα πάει στην Ολομέλεια, θα παραμείνει σε εκκρεμότητα με μια de facto πολιτική εντολή που πρέπει να ε, υιοθετηθεί και να επιβεβαιωθεί από το Νέο Κοινοβούλιο και την Νέα Επιτροπή ΕΚΟΝ. Και μάλιστα κατεπηγόντως. Αρχές Ιουλίου, με σκοπό στις 14 με 17 Ιουλίου να περάσει από την Ολομέλεια. Πάντα για το 2014 μιλάμε. Ε, ε, έκθεση του κύριου Λάγκεν θα παρουσιαστεί αμέσως μετά την ανταλλαγή απόψε. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον Υπουργό και αργότερα στο διοικητή της Κεντρικής Τραπέζης. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να περάσω στην πιο όμορφη γλώσσα του κόσμου, όπως γνωρίζω εγώ, στη μητρική μου τη Λιθουανική. Ε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, είναι μεγάλη μου τιμή που συμμετέχω σε αυτή τη συνεδρίαση. Βρίσκομαι εδώ για τρίτη φορά. Τις δύο πρώτες φορές ε, είχα παραστεί ως μέλος της ΕΚΟΦΗΝ, πρόεδρος μάλλον της ΕΚΟΦΗΝ. εκπροσωπώ ένα πολύ μικρό κομμάτι της Ευρώπης που είναι πολύ σημαντικό για μένα, είναι η Λιθουανία, η χώρα μου. Η Λιθουανία αφενός ε, κατάφερε να αποδείξει ότι είναι ισότιμο και αξιόπιστο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα κράτος μέλος ε, που ξέρει πώς να οργανώσει εργασίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έχουμε δει στη συνεδρία της ΕΚΟΦΗΝ και σήμερα θα σας αποδείξω ότι για άλλη μια φορά η Λιθουανία είναι ένα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα κράτος μέλος το οποίο ε, έχει προσχωρήσει, πρόκειται να προσχωρήσει στη νομισματική ένωση. Θα είναι λοιπόν η 17η χώρα που θα έχει το ευρώ ως εθνικό νόμισμα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη Λιθουανία και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μου με αυτό το βήμα επιθυμεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει δυνατότερη. Γι' αυτό το λόγο επιθυμούμε να προσχωρήσουμε στην Ευρωζώνη. Με έναν τρόπο ανοιχτό και αποφασιστικό ταυτόχρονα. Να σας παρουσιάσω κάποια δεδομένα Διάφορα στοιχεία διανεμήθηκαν πριν από την παρούσα συνεδρίαση, καθώς και διάφορα έγγραφα που φέραμε από το Βίλνιους, με κάποια σημαντικά σημεία, τα οποία καλό θα είναι να τονιστούν στη σημερινή συζήτηση. Η βασική ιδέα που θα ήθελα να σας παρουσιάσω είναι ότι επειδή κατά την άποψη μου η Λιθουανία είναι έτοιμη να υιοθετήσει το ευρώ και να προσχωρήσει στην ευρωζώνη, ε, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αυτή η προσχώρηση μόνο ως ωφέλη ε, αλλά και ως δεσμεύσεις για τη χώρα όπως ισχύει και για οποιαδήποτε χώρα της Ευρωζώνης η οποία Ευρωζώνη έχει διευρυνθεί πλέον αρκετά 18 χώρες εμείς προσπαθούμε τώρα να γίνουμε 19η πολλές δεσμεύσεις απορρέουν από την προσχώρηση στην Ευρωζώνη για ένα κράτος μέλος συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής ε, στο μηχανισμό σταθερότητας, ε, στην Τραπεζική Ένωση, ε, δραστηριότητες στις οποίες έχουμε συμμετάσχει ενεργά, αλλά και επιπλέον απαιτήσει επιτήρηση του προπολογισμού υπό το του ΠΑΚ, υιοθέτηση των διατάξεων του νομοθετικού συμφώνου και εγώ πρέπει να πω ειλικρινά ότι δεν έχουμε ακόμα ολοκλήρωση όλες τις εργασίες επί όλων αυτών των θεμάτων. Απομένουν πολλά να γίνουν Υπάρχουν συστάσεις συγκεκριμένες για κάθε χώρα. Υπάρχει σύσταση 1 που αφορά αυτόν ακριβώς το δημοσιονομικό τομέα. Ο δημοσιονομικός τομέας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί αυτός ο τομέας από εμά. Στη δημοσιονομική πολιτική η Λιθουανία έδειξε αυστηρότητα και παραγωγικότητα. Ξεκινήσαμε από 10% έλλειμμα το 2009 με ε, το εκτιμόμενο 2,5% το 2013. Αυτά είναι προκατακτικά στοιχεία, δεν είναι ακόμα στοιχεία της Eurostat. Έχουμε και δικά μας στοιχεία αργότερα πιο αξιόπιστα, αλλά αυτό αποτελεί απόδειξη ότι στα δημοσιονομικά μας δείχνουμε σύνεση η εμπιστοσύνη στις λιθουανικές πολιτικές επίσης αντικατοπτρίζεται ε, στα αρκετά χαμηλά επιτόκια. Όσον αφορά το μέλλον της χώρας μας, θεωρούμε ότι η υιοθέτηση του ευρώ δεν είναι το τελευταίο βήμα, δεν είναι το τελευταίο βαγόνι του τρένου, ούτε η τελευταία στάση του. Μετά από την προσχώρηση του ευρώ θα πρέπει να προετοιμαστούμε για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. Εκεί θα επισέλθουν τα κριτήρια του Μάστριχτ, ε, τα οποία δεν συνεπάγονται μορφώση μόνο με μια σειρά στοιχείων που προβλέπονται στις συνθήκες του Μάστρεκτ, αλλά ε, αναφέρονται και στην βιωσιμότητα. Θεωρώ ότι έχουμε αποδείξει τις προθέσεις μας ε, να υπάρξουμε βιώσιμοι στις παρουσίες πολιτικές μας. Επιδιώκουμε ενεργά μέτρα πολιτικής σε πολλούς, πολλοί αριθμούς τομείς οικονομικής ανάπτυξης. Έχουμε προβεί σε μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό τομέα. Θα τις βρείτε στα έγγραφα που σας έχουμε μοιράσει. Ένα από τα κυριότερα έργα για τη Λιθουανία είναι το ενεργειακό τερματικό που θα πρέπει να ολοκληρώσει ο ενεργειακός. Συγγνώμη, ο σταθμός ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα μας ε, ε, θα βοηθήσει να ενσωματώσουμε τα ενεργειακά μας συστήματα στα ευρωπαϊκά δίκτυα. αλλά και η ανακαίνιση των δημοσιοκτηρίων, η αναβάθμιση τους που θα επιλύσει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και το οποίο έχει αναφερθεί σε σχέδια εκθέσεων του, στο σχέδιο εκθέσεων του συναδέλφου Βέρνερ Λάγκεν αφορά την ενεργειακή απόδοση η οποία δεν βρίσκεται στα επίπεδα που θα επιθυμούσαμε. Δημιουργούμε επίσης ένα περιβάλλον ε, ε, φιλικό προς επιχείρηση στη Λιθουανία. Έχουμε προχωρήσει αρκετά βελτιώνοντας τη χωροταξία, τις διαδικασίες αφαιρεγγιότητας. Έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε την αφαιρεγγιότητα για ε, φυσικά πρόσωπα, το οποίο είναι κάτι καινούργιο στη Λιθουανία. Έχουμε κάνει τροπολογίες στον εργασιακό κώδικα, οι οποίες συζητώνται στο Κοινοβούλιο. Έτσι ελπίζουμε να γίνει πιο φιλικό προς επιχειρήσεις στο περιβάλλον της χώρας μας. Επίσης έχουμε κάνει κάποια βήματα διαρθρωτικά όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις της κοινωνικές δαπάνες. Έχουμε διαθέσει τα κοινωνικά ταμεία στους Δήμους ώστε να έχουν καλύτερο έλεγχο των καταβολών χρημάτων μόνο προς όσους τα χρειάζονται. Κάτι που απέδειξε την αποτελεσματικότητά του σε πέντε δήμους και επεκτείνουμε συνεπώς το σύστημα αυτό σε ολόκληρη την επικράτεια. Έχουν ληφθεί επίσης τελευταία μέτρα για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης. Και το τονίζω ήταν ε, μια σκληρή διαδικασία, αλλά δεν συμμορφώναστε ακόμα με τις απαιτήσει ε, ε, εισαγωγής νέων φόρων Είναι πολύ σημαντικό αυτό το φορολογικό κομμάτι για μας και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την εισπράξη Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θεωρούμε ότι οι προοπτικές Λιθουανίας είναι καλές στην Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη θα μας είναι ιδιαίτερα επωφελής, θα βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα, θα ενισχύσει την οικονομική μας ανάπτυξη και τέλος θα επιτύχει τον τελικό μας στόχο να βελτιώσουμε τις ζωές των πολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Πρόεδρε, ίσως μπορούμε τώρα να δώσουμε το λόγο στον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας να μας παρουσιάσει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, ε, ο διοικητής της Τράπεζας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, εκτιμώ αυτήν την ευκαιρία να σας ενημερώσω σχετικά με την κατάσταση της λιθουανικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση θα συμβάλλει στην διαμόρφωση μιας εικόνας. Θα επικεντρωθώ στα θέματα τα οποία συνδέονται στενά με την εντολή της Κεντρικής Τράπεζας. Καταρχάς δηλαδή, πώς αντιμετώπισε η λιθουανική οικονομία την κρίση. Δεύτερον, πώς βλέπουμε την ε, σταθερότητα των τιμών, διότι αυτό είναι θέμα που εμπίπτει στην εντολή της Κεντρικής Τράπεζας και τρίτον, ε, πώς είναι τα πράγματα στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η λιθουανική οικονομία ανέκαμψε μετά την κρίση και επιδεικνύει ανάπτυξη. Η... Φέτος θα ξεπεράσουμε τα επίπεδα παραγωγής πριν την κρίση και η συσσωρευτική αύξηση του ΑΕΠ από το 2009 και μετά ε, ξεπερνάει το 15%. Τα βασικά στοιχεία της ε, στρατηγικής ε, προσαρμογής ήταν η πολιτική ανταπόκριση, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η οικονομική ευελιξία. Η αποκατάσταση της ε, ισορροπίας έχει επιτευχθεί με την ε, ευελιξία στην ε, αγορά εργασίας και την αγορά προϊόντων. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν ισοσκελισμένους λογαριασμούς. Η ανταγωνιστικότητα έχει βελτιωθεί με σημαντικές προσαρμογές στο κόστος εργασίας ανατεμάχιο παραγωγής. Η οικονομική ανάκαψη φάνηκε κυρίως ε, στο εμπόριο, έχει σταθεροποιηθεί και η εγχώρια ζήτηση. Οι πραγματικές εξαγωγές ξεπερνούν κατά 40% το υψηλότερο σημείο που είχαν φτάσει πριν την κρίση και η ανεργία έχει πέσει σχεδόν στο μισό από την υψηλότερη τιμή της κρίσης και αυτή τη στιγμή βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο της ε, περιοχής του ευρώ της ζώνης του ευρώ. Η διαδικασία προσαρμογής είναι αρκετά ευέλικτη και μπορούμε έτσι να προσαρμοζόμαστε στις, ε, να προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας όποτε είναι απαραίτητο αυτό. Η πίεση στις εγχώριες τιμές έχει περιοριστεί και ο πληθωρισμός βρίσκεται κάτω από το κριτήριο σταθερότητας των τιμών. Ο μέσος πληθωρισμός αναμένεται να περιοριστεί στο 0,7% το πρώτο τρίμηνο του 2014. Όσον αφορά την ε, βιωσιμότητα σε μεσοπρόθεσμο στάδιο, οι προβλέψεις είναι ενθαρρυντικές. Η πρόληψη κακών εξελίξεων θα ε, αντισταθμιστεί με ε, εργαλεία μακροπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή οι κλειδονισμοί στις ε, τιμές στην Λιθουανία ήταν αρκετά ισχυρές λόγω του υψηλού ποσοστού τιμών τροφίμων και αγαθών στο καλάθι του καταναλωτή. Ωστόσο, οι κλειδονισμοί αυτοί έχουν περιοριστεί και επίσης έχουμε αυτή τη στιγμή πολιτικές οι οποίες θα μειώσουν ε, την ε, χρήση ενέργειας και από την άλλη θα έχουμε και διαφοροποίηση στις ενεργειακές τιμές. Οι πρωτοβουλίες αυτές, όπως είναι η ε, ανακαίνιση σπιτιών, ο σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο διαχωρισμός των δικτύων παροχής και διανομής του αερίου, ε, στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος ε, να πω λίγα λόγια για τον χρηματοπιστωτικό μας τομέα. Ενώ υπάρχουν κριτήρια σύγκλησης για να ε, εντοπιστούν τα προβλήματα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η κρίση μας θύμισε ότι υπάρχουν σημαντικές διασυνδέσεις ανάμεσα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την πραγματική οικονομία. Κατά την αξιολόγηση της ε, σύγκλησης και της οικονομικής ε, βιωσιμότητας ε, έχουμε πολλά να πούμε όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας λοιπόν στην Λιθουανία δεσπόζεται από, την, από τον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα, ο οποίος δεν είναι υπερβολικό σε μέγεθο και οι τράπεζε αντιπροσωπεύουν το 65% του ΑΕΠ. Οι χρηματοδοτικές δομές ε, έχουν κυρίως προσανατολισμό το εσωτερικό της χώρας και οι τράπεζες ε, έχουν αναλογία ε, χρεών και καταθέσεων που ανέρχεται σε 107%. Επίσης, οι καταθέσεις αλλοδαπών είναι αμελητές το 3%. Ο τραπεζικός τομέας έχει πάνω από το διπλάσιο κεφάλαιο από αυτό που απαιτείται από την ε, Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας και τα κεφάλαια αυτά είναι υψηλής ποιότητας. Το 99% ε, ανήκουν ε, στη ζώνη 1, Tier 1. Και επίσης τα κακά χρέη έχουν μειωθεί και αυτή τη στιγμή περιορίζονται στο 10,7%. οι συνθήκες ε, δανεισμού έχουν εξομαλυθεί και δεν υπάρχει υπερβολικό χρέος. Επίσης, ε, ε, τα χρέη των νοικοκυριών είναι τα δεύτερα πιο χαμηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 43,1% του ονομαστικού ΑΕΠ. το χαρτοφυλάκιο δανεισμού ε, αναμένεται να αυξηθεί κατά 3% το 2014 και οι ε, έρευνες της ε, Τράπεζας της Λιθουανίας δεν δείχνουν να υπάρχουν δανειστικοί περιορισμοί. Επίσης έχουμε ένα κουτί εργαλείων για να αποφύγουμε τα μη βιώσιμα χρέη και Η Τράπεζα της ε, Λιθουανίας ως εποπτική αρχή είναι διατεθειμένη να ε, προσχωρήσει στον ε, ενιαίο εποπτικό μηχανισμό με την προσχώρηση της χώρας στην ζώνη του ευρώ. Όπως έχει σημειωθεί, ο χρηματοπιστωτικός τομέας βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θα κλείσω εδώ και ευχαρίστως θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δίκητα, έχουμε δύο μιλητές και παρακαλώ τα μέλη που θα κάνουν ερωτήσεις τώρα να ξεκαθαρίσουν σε ποιον απευθύνουν την ερώτηση. Επίσης, παρακαλείστε να μοιράσετε τις απαντήσεις οι δυο σας για να μην έχουμε επικαλύψεις. Αρχίζουμε αμέσως με τον εισηγητή μας, τον κύριο Λάγκεν. Okay, Ωραία, ευχαριστώ πολύ θα ήθελα να πω καταρχάς ότι χαίρομαι που έκανε αίτηση η Λιθουανία να προσχωρήσει στη ζώνη του ευρώ. Είναι χαρμόσυνο πραγματικά. Πριν από μία διετία γινόντουσαν μεγάλες συζητήσεις εάν μπορεί στο διενικές να επιζήσει η Ευρωζώνη. Από το 2012 και μετά αυτά είναι παρελθόν. Και κάθε νέο μέλος το δεχόμαστε με ανοιχτές αγκάλες. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά θα κάνω αυτή τη σύσταση. Αυτό θα το πούμε στο τέλος όμως και θα το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρουσιάσεις σας. Είδα και την τελευταία, την πιο πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου των αρχών Μαρτίου. Είναι εξαιρετικά θετική. Η Λιθουανία είχε κάποιους στόχους για απρόσκοπτη προσχώρηση στο ευρώ τους έχει καλύψει σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια οριστικούς αριθμούς δεν έχουμε ακόμα και δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε και τελεσίδικα. Απλώς να κάνω λοιπόν μερικές ερωτήσεις. Ε, πρώτον, ε, πώς ξεπεράσατε την κρίση στις χρηματαγορές. Εξ όσων γνωρίζω και αν δεν απατώμε το 2009 η Λιθουανία είχε ε, τεράστια μείωση ε, ε, του ΑΕΠ κατά 14,8 παρακαλώ Πολύ γρήγορα όμως το κάλυψε αυτό το κενό. Ταυτόχρονα ε, μεταξύ μισθών και παραγωγικότητας υπήρχε μεγάλη απόσταση, μεγάλο χάσμα που παρατηρήθηκε και στη νέα Ευρω... νότια συγγνώμη, Ευρώπη ως μεγάλο πρόβλημα και αυτό το κάλυψε η Λιθουανία. Τι κάνατε συγκεκριμένα στη χώρα σας, έτσι ε, ώστε να καλύψετε αυτά τα κενά και πού οφείλεται καν αυτό το κενό και το χάσμα που παρατηρήθηκε. Ήταν η πρώτη μου ερώτηση αυτή. Και η δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο διοικητή της ε, Κεντρικής Τραπέζης. το τραπεζικό σύστημα, ο κλάδος ο τραπεζικός, δεν μου αρέσει να το ονομάζω βιομηχανία γιατί έχουν γίνει πολλές ανοησίες εκεί. Ε, ο κλάδος ε, ή ο δικός σας ο τραπεζικός εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από σκανδιναβικές τράπεζες. Πώς φαντάζεστε την πορεία, ειδικά μιλώ εδώ για τις σουηδικές τράπεζες, θα συνδεθούν στην είσοδο του ευρώ, διότι μέχρι τώρα η Σουηδία δεν είναι μέλος του ευρώ, λόγω πολιτικής απόφασης παρόλο που πληρεί τα κριτήρια και που κανονικά θα όφιλε, διότι είναι μια χώρα ε, που έχει εξαίρεση η ε, πολιτική απόφαση μέχρι τώρα ήταν διαφορετική. Αλλά εκεί υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα με τις σκανδιναβικές τράπεζες που κυριαρχούν στη Λιθωνία. Η πρώτη μου ερώτηση απευθυνόταν προς τον Υπουργό και η δεύτερη στον κυβερνήτη, το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Παρακαλώ να απαντήσει πρώτα ο διοικητής της Τραπέζης. Ευχαριστώ Βερνέρ για αυτή την πολύ σημαντική ερώτηση. Η κατάσταση με τις αμοιβέ ε, στην αγορά εργασίας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για τον πολύ απλό λόγο ότι εξακολουθούμε να θεωρούμε τη χώρα μας ως μια χώρα φθηνών εργατικών. Αρκετά φθηνών μπορεί να θεωρηθεί. Φυσικά υπάρχουν χώρες στον κόσμο με πολύ χαμηλότερες αμοιβέ. Αλλά δεδομένου του υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης που κληρονομήσαμε από τα παλιότερα χρόνια. Ε, υπάρχουν διάφορα πολύ θετικά χαρακτηριστικά στο εργατικό μας δυναμικό και μας ενδιαφέρει να αξιοποιήσουμε αυτό το εργατικό δυναμικό με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Είχαμε ανεξέλεγκτη αύξηση των αμοιβών πριν από την κρίση, πριν το 2008. Μερικές φορές ε, η αύξηση ήταν ε, διψήφια. Λίγο χαμηλότερη βέβαια από κάποιες γειτονικές χώρες. Αλλά παρόλα αυτά ήταν αρκετά υψηλή η αύξηση αυτή. Μετά είχαμε εσωτερική υποτίμηση, η οποία ήταν επώδυνη Λόγω της σημερινής μας σύνδεσης με το ευρώ έχουμε συνδέσει από τις 2 Φεβρουαρίου του 2012 το νομισμά μας με το ευρώ. Πριν από αυτό ήταν συνδεδεμένο με το δολάριο. Για δύο δεκαετίες λοιπόν αυτή η σύνδεση ήταν ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για μια τόσο μικρή χώρα, με τόσο μικρή οικονομία. Και μας επέτρεψε να μην ολιστήσουμε, αλλά από την άλλη δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να μειώσουμε τις αμοιβέ και τους μισθούς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Φυσικά στο δημόσιο τομέα έχουμε κάποιες εκκρεμείς ε, αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν αυτές οι περικοπές στους μισθούς και πιστεύω ότι μας συμφέρει στην Ευρωζώνη, στην Ευρώπη και με χώρες που έχουν παρόμοια νομισματική σύνδεση να έχουμε κάποια τεχνογνωσία, κάποιο εγχειρίδιο το οποίο θα μας λέει πώς να προχωράμε με την εσωτερική υποτίμηση και τη μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, στο, δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα έγινε μια προσαρμογή ιδίω ταχυτήτων. Κάποιες ε, επιχειρήσεις απέλησαν και αυξήθηκε έτσι και η μετανάστευση από τη Λιθουανία. Σε άλλες επιχειρήσεις όμως αποφάσισαν να περικόψουν τους μισθούς όλων. Και αυτές τελικά οι επιχειρήσεις είναι αυτές που υπήρξαν πιο αποτελεσματικές και είναι πιο ε, αποδοτικές και υγιείς σήμερα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το μάθημα που, το δίδαγμα που αποκόμισαν οι λιθουανικές επιχειρήσεις. Εξαιρετικό μάθημα. Ε, η κρίση είναι ακόμα κάτι που θυμόμαστε καλά πολύ φρέσκο. Μέχρι να την ξεχάσουμε θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να υλοποιήσουμε βέλτιστες πρακτικές ε, ε, που έχουμε δει τόσο σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις. όσο και στι γειτονικέ χώρε τη Λιθουανία. Εμεί τώρα προβλέπουμε 5-6% ονομαστική ε, αύξηση των μισθών των εργαζομένων τη Λιθουανία και στου δύο που θα πρέπει λογικά να συνοδευτεί με αύξηση της παραγωγικότητας. Αλλά πιστεύω ότι και εδώ ο δημόσιος τομέας πρέπει να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση της παραγωγής δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες, καλύτερης εκπαίδευσης των ανθρώπων, όχι μόνο στη Λιθανία, σε ολόκληρη την Ευρώπη η υιοθέτηση του ευρώ θα αποτελέσει ακόμα έναν συντελεστή, όχι τον κύριο, αλλά έναν από του συντελεστέ που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτίωση τη κατάσταση στην αγορά εργασία. Και ε, να βοηθήσουν και σε αυτή τη σύγκληση των εισοδημάτων των, του πληθυσμού μα με τον Ευρωπαϊκό μεσόωρο. Ευχαριστώ. Ε, έχουμε ενδιαφέρουσα ε, κατάσταση, λέει ο κύριος Βασιλιάουσκας, διοικητής της ε, Κεντρικής Τράπεζας, ε, με, όπως σας είπα, θηγατρικές σκανδιναβικών τραπεζών, όπως σας είπα, 90% των τραπεζών μας έχουν ιδιοκτησιακό καθεστώς σκανδιναβικής τράπεζας, είναι υποκαταστήματα ή θηγατρικές. Και οι τρεις μεγαλύτερες, αν μπούμε στην Ευρωζώνη, αυτομάτως δηλαδή, αν είμαστε τμήμα του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, ε, θα είναι υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρέπει όμως να σας πω ότι έχουμε πολύ καλή εμπειρία συνεργασίας ε, με τη Λιθουανική Εποπτική ε, Αρχή της Λιθουανίας και των Σκανδιναβικών χωρών, ιδιαίτερα της Σουηδίας. Κατά την παρελθούσα δεκαετία, ας πούμε, ήταν μοναδική η συνεργασία μας, πραγματικά υπόδειγμα. Ε, ήταν βορή ευρωπαϊκού τύπου, βαλτικού τύπου εποπτεία. Τι σημαίνει αυτό, ότι ε, παρακολουθούμε και ελέγχουμε από κοινού και στη συνεργασία με τους Σουηδούς συναδέλφους στις τράπεζές μας. Τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή συνταχθούμε στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Θα συνεχίσουμε αυτό το πρότυπο συνεργασίας και το μοντέλο βεβαίως. Συμμετέχουν εκεί ε, από εκείνη τη στιγμή και της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Πέντε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Χαίρομαι που υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τηρούν τις συμφωνίες και τις υποχρεώσεις τους παρά τις δυσκολίες που συναντούν. Η Λιθουανία ε, πληρούσε σχεδόν τα κριτήρια του ευρώ το 2007. Στο μεταξύ όμως ήρθε η οικονομική κρίση Η Λιθουανία ξεπέρασε τα προβλήματα και χαίρομαι πάρα πολύ που η Λιθουανία είναι πια έτοιμη να προσχωρήσει στο ευρώ και που σύντομα και τα τρία κράτη της Βαλτικής θα είναι μέλη της ζώνης του ευρώ. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το πώς βλέπουν οι απλοί άνθρωποι στη Λιθουανία τα σχέδια αυτά. Το κοινό της Λιθουανίας τι λέει για όλα αυτά και έχετε σκεφτεί τον κίνδυνο αύξησης των τιμών. Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για να αποφύγετε τις αυξήσεις. Στην Εστονία και τη Λετονία υπάρχει και μια πτυχή πολιτικής ασφαλείας όσον αφορά την υιοθέτηση του ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν συμβεί στην ε, Ουκρανία, νομίζω ότι ο ενθουσιασμός των Λιθουανών ε, θα είναι μεγαλύτερος όταν μιλάμε για την ε, υιοθέτηση του ευρώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για όλη τη δουλειά που έχετε κάνει. Οι σοσιαλδημοκράτες στηρίζουν τις προσπάθειές σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παντάρ για τα καλά σας λόγια τα οποία απευθύνεται στους γειτόνους σας. Είναι πολύ σημαντικό οι τρεις χώρες της Βαλτικής που αποτελούν ε, μια ενιαία οικονομική υποπεριοχή, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οικονομική περιοχή. Μιλάμε λοιπόν για μια υποπεριοχή η οποία θα προσχωρήσει στην ε, Ευρωζώνη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένας από τους λόγους που θέλουμε να προσχωρήσουμε στη ζώνη του ευρώ όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όσον αφορά τις ερωτήσεις σας, οι απόψει των απλών ανθρώπων είναι ανάλογε με αυτόν σε όλες τις χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωζώνη μετά τη δημιουργία της. Είναι επιφυλακτική. Νομίζω όμω ότι μπορούμε να... Ε, ιστορία επιτυχίε της Εστονία που το 2011-2012 είχε 40-45% των ανθρώπων υπέρ ε, του ευρώ, τώρα όμως ε, στο τέλος του 2013 το 78% είναι υπέρ του ευρώ στην Εστονία. Η Εστονία λοιπόν ήδη ε, έχει δει τους καρπούς ε, της υιοθέτηση του ευρώ και αυτό είναι καλό παράδειγμα για τη Λετωνία και για μας ε, και θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την επιφύλαξη όχι με προπαγάνδα αλλά με εκστρατείες πληροφόρησης τις οποίες ήδη έχουμε ξεκινήσει και που θα συνεχιστούν και στο δεύτερο εξάμεινο αυτού του έτους. Πιστεύω ότι έτσι θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την ε, θέση του κόσμου απέναντι στο ευρώ. Υπάρχει ο κίνδυνος της αύξησης ε, των τιμών. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε μια γειτονική χώρα που εισήγαγε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου φέτος, έτσι μπορούμε ήδη να παρατηρήσουμε εάν έχουν ε, αυξηθεί οι τιμές. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πραγματικό παράδειγμα το οποίο μπορούμε να δείξουμε στους ανθρώπους. Μπορούν να πάνε στη Λιτωνία διότι δεν ε, έχουμε πια εσωτερικά σύνορα στην Ευρώπη. Θα δημιουργηθεί όμως ένα σύστημα ελέγχου. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα ε, κρατικών θεσμικών ε, οργάνων. Συμμετέχουν όμως και κάποιες ενώσεις κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, και έχουμε διαθέσει κονδύλια για την επιστροφή των δαπανών αυτών ε, των οργανώσεων, ώστε να δημιουργήσουμε αυστηρούς ελέγχους για την δίκαιη παρακολούθηση των τιμών. Δεν θα εμποδίσουμε τις εξελίξεις στις τιμές, διότι αυτό οικονομικά δεν θα ήταν έξυπνο. Δεν μπορεί να σταματήσει κανείς τις εξελίξεις των τιμών, διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη των τιμών αργότερα. Δεν θέλουμε να έχουμε αρνητικές εξελίξεις στον τομέα των τιμών. Θα τις αφήσουμε να εξελιχθούν με φυσικό τρόπο, αλλά τα συστήματα θα πρέπει να προσαρμοστούν στις τιμές με το νέο νόμισμα. Και προς τον σκοπό αυτό θα επιβάλλουμε την ε, διπλή αναγραφή των τιμών και στα δύο νομίσματα δηλαδή ε, έξι μήνες πριν την εισαγωγή του ευρώ, ξεκινάμε φέτος το καλοκαίρι και θα συνεχιστεί αυτό και έξι μήνες μετά την εισαγωγή του ευρώ. Πιστεύουμε ότι αυτό θα αρκέσει και επίσης ε, όσον αφορά την τελευταία ερώτηση του κυρίου Παντάρ. Δεν θα ήθελα να πω ότι θα εκμεταλλευτούμε την κατάσταση της Ουκρανίας απλά για να βελτιώσουμε την στάση του κόσμου απέναντι στο ευρώ, αλλά Νομίζω ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα στην κεντρική Ευρώπη θα αναγκάσει τον κόσμο να σκεφτεί πού ζούμε, ποια είναι η ιστορία μας, ποιες είναι οι φιλοδοξίες μας, οι αξίες μας και ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κύριε Διοικητά. Ναι, ευχαριστώ. Ε, σε σχέση με τον πληθωρισμό να πω κάτι μόνο. 0,7% είναι η αύξηση του ε, προϋπολογισμού ετήσια για φέτος και ενδεχομένως σύμφωνα με τα στοιχεία μας για το 2015 ο πληθωρισμός μπορεί να είναι της τάξεως του 1,5% μέχρι 1,9% το 2016. Κάπου εκεί δηλαδή κειμενόμεθα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλούμε για ε, πιθανή εκτόξευση των τιμών στη Λιθουανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος, και εξ ονόματος των Φιλελευθέρων, ο κύριος Τρεμόσα, παρακαλώ. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αρχές της ε, Λιθουανίας ε, για την παρουσία τους εδώ και είμαι ικανοποιημένος πρέπει να πω που υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουν να μπουν στο ευρώ. Διότι γνωρίζουμε ότι η Ευρωζώνη δεν είναι κανένα ιδεατός κόσμος αλλά ενισχύει εν πάση περιπτώσει την ε, στράτευσή μας και τη δική μας προσήλωση και μπορούμε να γυρνάμε στις χώρες μας και να λέμε ότι ορίστε υπάρχουν χώρες που αγωνίζονται και κάνουν σκληρές θυσίες για να μπουν στο ευρώ, στο κοινό μας νόμισμα. Μια ερώτηση έχω μόνο. Θα ήθελα παρακαλώ να μάθω ποια είναι η άποψή σας για την Τραπεζική Ένωση όπως έχει σχεδιαστεί αυτό τον καιρό. Διότι όπως ακούστηκε, οι σκανδιναβικές τράπεζες έχουν πολύ ισχυρή παρουσία στη χώρα σας και θα ήθελα παρακαλώ την άποψή σας γι' αυτό και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση, αν μπορεί να βελτιωθεί και αν θα είναι σε άνετη θέση μια χώρα να είναι στο ευρώ και να εξαρτάται τόσο πολύ ο τραπεζικό τομέα τη από τη Σουηδία. Ιδιαίτερα γιατί γίνεται και συζήτηση για αυτά τα θέματα. Αυτά. Α, και μια άλλη ερώτηση. Θα ήθελα επίσης να μάθω εάν ε, ε, η Λιθουανία εφαρμόζει το δημοσιονομικό σύμφωνο και το λεγόμενο χρυσό κανόνα περί ισοσκελισμένων προϋπολογισμών για να αποφευθούν ε, κάποια αρνητικά φαινόμενα στο μέλλον. Ποια είναι η πρακτική και η βέλτιστη εμπειρία σας. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Με τη σειρά θα απαντήσω. Τραπεζική Ένωση πρώτα απ' όλα. Ήμουν παρόν όταν γεννήθηκε αυτός ο συμβιβασμός της 18 Δεκεμβρίου πέρυσι στο Συμβούλιο Κοφίν, το οποίο προέδρευα εκείνη τη στιγμή. Ήταν ένας δύσκολος συμβιβασμός, αλλά έγινε με συνένεση. Αυτό λέει πολλά. Τώρα ξέρω ότι οι τριμερείς διάλογοι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αρκετά δύσκολη. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι για μένα η διαδικασία δημιουργίας ενός ε, ενιαίου μηχανισμού εποπτείας είναι μια μοναδική διαδικασία στην ιστορία της Ευρώπης. Είναι ο πρώτος μηχανισμός στο είδος του. Διότι ήδη κάποιες φορές είχαμε αυτό που ονομαζόταν Eurogroup Plus, όπου οι υπουργοί του Eurogroup ε, ε, συμμετείχαν, καθώς και οι υπουργοί χωρών που δεν ανήκαν στο Eurogroup αλλά και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συζητούσαν διακυβερνητικές συμφωνίες που γνωρίζω ότι δημιουργούν πολλές αμφιβολίες για, σε κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά που επίσημα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αποφασίζουν οι υπουργοί και οι κυβέρνηση. Η γενικότερη άτυπη άποψη είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι αυτή η διάρθρωση δύο πυλώνων του ενιαίου ε, ε, μηχανισμού εξυγίανσης ε, που είναι το μόνο που λείπει στο οικοδόμημα της Τραπεζικής Ένωσης θα λειτουργήσει. Και θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε με εσάς, με τους υπουργούς, μεταξύ των υπουργών και ε, του μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχοντας την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σωστή, τρίτου συμμετέχοντας στους τριμερείς ε, διαλόγους. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε κάτι το οποίο θα είναι υποφελές για όλα τα κράτη-μέλη και την ενιαία αγορά, αλλά και τους λαούς της Ευρώπης. Όσον αφορά το δημοσιονομικό σύμφωνο, βρισκόμαστε σε φάση προετοιμασίας ε, της νομοθεσίας που θα εφαρμόσει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και που θα το ενσωματώσει στη Λιθουανική νομοθεσία. Έχουμε ήδη μία πράξη δημοσιονομικής πειθαρχίας που υιοθετήθηκε το 2007, ωστόσο, που εισήγαγε κάποιους νέους θευματουργούς κανόνες ελέγχου της αύξησης των δημοσιονομικών δαπανών. Αυτή ο όμως πιστεύω βοήθησε πάρα πολύ, πολύ αποτελεσματικά να επιτύχουμε αυτή την τάση του δημοσιονομικού ελλείμματος που βλέπετε στα φύλλα τα οποία σας δώσαμε, που σας μοιράσαμε. Από 9% το 2009 μειώθηκε στο 2,9% και σε ίσως ως προπολογισμό το 2016. Φυσικά απομένουν πολλά να γίνουν σε αυτόν τον τομέα. Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε ένα ιδιαίτερο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο για τα δημόσια οικονομικά. Η μη ύπαρξή δεν είναι κάτι που εγκυμονεί κινδύνους, αλλά βοηθάει στην αποφυγή απρόβλεπτων αποτελεσμάτων στο τέλος του έτους. Και η δημοσιονομική πειθαρχία θα έχει εφαρμοστεί στους Δήμους το φθινόπωρο φέτο. και ο προϋπολογισμός του 2015 θα βασίζεται σε αυτούς τους κανόνες. Το δημοσιονομικό σύμφωνο θα ενσωματωθεί στη λιθανική νομοθεσία φυσικά φέτος πριν μπούμε στην Ευρωζώνη. Διότι είναι κάτι απολύτω αναγκαίο. Ο διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να προσθέσει κάτι για την Τραπεζική Ένωση και τι Σουηδικέ Τράπεζε. Ε, ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε πιστεύω με το σημερινό μοντέλο συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής, Εποπτικής Αρχής και της Σουηδικής ε, Εποπτικής Αρχής ή υπό την ηγεσία των ομάδων του της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό το μοντέλο λειτουργεί στη δική μας περίπτωση. Μπορούμε λοιπόν να το συνεχίσουμε. E ευχαριστώ εκ μέρους του ECR. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπόκερς. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους ε, των Ευρωπαίων ε, Συντηρητικών θα ήθελα να ε, εκφράσω την εκτίμησή μας στην Λιθουανία για τις μεγάλες θυσίες που έχει κάνει, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά θα έλεγα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ετών, για να απαλλαγούν από την κληρονομιά της Σοβιετικής Ένωσης. Η προσαρμογή και μετάβαση των ε, χωρών της Βαλτικής ήταν πολύ πιο δύσκολη από ότι στην ε, κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Εγώ είμαι ε, Ούγγρος. Θα γνωρίζετε ότι οι χώρες του Βίσιγκραντ είχαν καλύτερη ε, τύχη, όχι όλες, αλλά ε, κάποιες από αυτές. Ε, θα ήθελα λοιπόν να επενέσω τα όσα, έχουν, τα όσα έχει καταφέρει όχι μόνο η Λιθουανία, αλλά και οι άλλες δύο χώρες της Βαλτικής τα τελευταία 24 χρόνια. Μία πτυχή την οποία θα πρέπει να τονίσουμε έχει να κάνει με το Συμβούλιο Συναλλάγματος. Είναι, είναι ένας ε, κορσές. Ε, όλοι γνωρίζουμε ότι Όταν ε, ασκείται έτσι η νομισματική κυριαρχία, τότε οι περισσότεροι περιορισμοί επιβάλλονται στην εργασιακή πολιτική κλπ. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η διατήρηση αυτής της ρύθμισης για τόσο καιρό χωρίς προβλήματα είναι σημαντικό επίτευγμα και ξεπερνάει κατά πολύ τις ε, συνέπειες της κρίσης. Όλη η Ευρωζώνη ε, μπορεί να μάθει κάτι σημαντικό από αυτό. Η Λιθουανία όπως και η Λετωνία και η Εστονία είχαν το θάρρος ε, να ε, υποτιμήσουν το νόμισμά τους όταν ήταν αυτό απαραίτητο, όταν πια δεν ήταν βιώσιμο το μισθολογικό κόστος και δεν ακολουθούσε την παραγωγικότητα πριν την κρίση. Μία χώρα λοιπόν που κατάφερε να κάνει κάτι τέτοιο πριν προσχωρήσει στη ζώνη του ευρώ, διότι υπάρχουν χώρες εντός της Ευρωζώνης που δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό μάθημα για όλους μας και θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου. Έχω την εξή ερώτηση. Θα μου επιτρέψετε να επενέσω τα όσα έχει γράψει στην έκθεσή του ο Βέρνερ. Μία μικρή έκθεση μόνο ή μία πρόταση θα έλεγα που έχει να κάνει με την ε, εξωτερική ισορροπία. Αναφέρομαι ε, στο τρέχον ισοζύγιο και στο εξωτερικό χρέος. Είδαμε ότι αυτά είναι σημαντικά, διότι παλιότερα ένιωθε κανείς ότι σε μια νομισματική ε, ένωση αυτό είναι απλά ένα στατιστικό νούμερο, αλλά δεν είναι. Βλέπουμε τώρα ότι η Λιθουανία μπορεί να αποφύγει και το μεγάλο έλλειμμα και το μεγάλο εξωτερικό έλλειμμα και το μεγάλο δημοσιονομικό και το μεγάλο εξωτερικό έλλειμμα. Δεν υπάρχει λοιπόν διπλό έλλειμμα ούτε διπλό χρέος αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να επανέλθει. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το έλλειμμα είναι χαμηλό επειδή δεν είναι και τόσο μεγάλη η ανάπτυξη και η Λιθουανία θα πρέπει να καλύψει τη διαφορά. Χρειάζεται επιπλέον επενδύσεις. Αν και όταν αυξηθούν οι επενδύσεις, μπορεί να δούμε και μεγαλύτερο ε, έλλειμμα. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτείτε πώς θέλετε να διαχειριστείτε το χρέος. Ευχαριστώ. Κύριε Μπρόκας, ε, κλέψατε σχεδόν όλο το χρόνο για τις ερωτήσεις. Ε, θα εκτιμούσα λοιπόν αν ο διοικητής και ο Υπουργός μπορούν να είναι σύντομοι στις απαντήσεις τους. Ε, εάν ο, ο εισηγητής ζητήσει εξαίρεση, ο πρόεδρος θα το δεχτεί. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Θα προσπαθήσω να απαντήσω αυτήν την όχι πολύ εύκολη ερώτηση. Βρισκόμαστε τώρα σε άλλη διάσταση από ό,τι βρισκόμασταν το 2008 πριν την κρίση και όσον αφορά την ε, διαχείριση ε, ε, σε περίπτωση που έχουμε φούσκες στο μέλλον, αυτό απαιτεί μακροπρόθεσμα μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να μπορέσει να αντιδράσει γρήγορα σε οποιαδήποτε αλλαγή στην οικονομία και ιδιαίτερα σε αλλαγές στην αγορά ακινήτων μας. Όπως είπα, στην Λιθουανία έχουμε δεσμευτικούς ε, κανόνες ε, όσον αφορά τις ε, αναλογίες χρέους εισοδήματος και την απόσβεση των χρεών. Αυτή τη στιγμή συζητάμε με το, συζητάμε στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο τη δυνατότητα διεύρυνσης της μακροπροληπτικής εντολής και στις ε, κοινοβουλευτικές αυτές ε, συζητήσεις. Συζητιέται η ύπαρξη νέου νόμου που να δίνει νέες αρμοδιότητες ε, στην κεντρική τράπεζα. Όλα αυτά τα εργαλεία θα μας βοηθήσουν να αποφύγουμε τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει να προσθέσει τίποτα ο υπουργό, οπότε πάμε μέσω στου πρασίνου και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπεσέτ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά, καλώ ορίσατε κυρίω η χώρα σα θα έλεγα. Χαιρόμαστε που ε, βαίνουν ε, καλώς τα πράγματα, είναι θετικές οι εξελίξεις και τα κριτήρια για την ένταξη της χώρας σας στην Ευρωζώνη είναι θετικά. Και πάνω απ' όλα χαιρόμαστε που έχετε και τέτοια πολιτική βούληση ε, ένταξη στην Ευρωζώνη. Που δεν είναι καθόλου υποζώνη, μάλλον υπερζώνη είναι στη ε, υπόθεση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Και χαιρόμαστε που έχετε και τόσο θετικό πνεύμα και αισιοδοξία ε, σε μια στιγμή που το Ουκρανικό κυριαρχεί και βαραίνει πάρα πολύ την όλη γενικότερη περιοχή. Ε, θα ήθελα να σας κάνω σύντομα τις εξής ερωτήσεις. Πρώτον, σύμφωνα και με τους προηγούμενους συναδέλφους του ΕΛΚ και των φιλελευθέρων, για την εξάρτηση του τραπεζικού σας τομέα από τις Σουηδικές τράπεζες και σκανδιναβικές γενικότερα. Απαντήσατε κύριε Δικητά, εξαίροντας ε, το μοντέλο συνεργασίας που έχετε με τη Σουηδική Εποπτική Αρχή, δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό αρκεί για να μας καθησυχάσει ως προς την ε, εύθραυστη ε, αυτή η υπερβολική εξάρτηση που έχουν οι τράπεζες σας από τις Σουηδικές τράπεζες. Και υπάρχει μία αντίφαση, έτσι, εξορισμού. Εντάσσεστε σε μια ζώνη νομισματική ε, με κυρίαρχες τράπεζες μιας χώρας που δεν ανήκει σε αυτή τη ζώνη. Ε, πώς εργάζεται για ένα ε, σύστημα έτσι πιο βιώσιμο και πιο καθησυχαστικό. Το δεύτερο, το φορολογικό σας σύστημα. Έχετε ένα ενιαίο φορολογικό συντελεστή, το λεγόμενο flat tax και για το φόρο εισοδήματος. Ε, αυτό δεν παράγει μόνο κοινωνική ανισότητα, αλλά δεν είναι και βιώσιμο μακροπρόθεσμο σε σχέση με ε, τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και τα δημόσια οικονομικά. Έχετε σκεφτεί σταδιακά και βαθμία να προχωρήσετε προς ε, ένα προοδευτικό φόρο εισοδήματος με αυξανόμενους προοδευτικά συντελεστές. Και μια τρίτη ερώτηση, αφού θα μπείτε στην Ευρωζώνη, πράγμα που σας εύχομαι και χαίρομαι γι' αυτό, ε, πώς σκέφτεστε από πλευρά σας να αντιμετωπίσετε ε, τα μεγάλα διακυβεύματα της Ευρωζώνης. Με ποια διακυβέρνηση, πώς τη φαντάζεστε τη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Ξέρετε ότι γίνεται μια ευρύτατη συζήτηση. Είστε υπέρ ενός ειδικού προπολογισμού για την Ευρωζώνη ξεχωριστού είστε υπέρ ε, μηχανισμού ε, σταδιακής συνένωση των ε, κρατικών χρεών. Ευχαριστώ, Υπουργό. Thank you for your question. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Την ερώτησή σας για τις σχέσεις του τραπεζικού τομέα θα τις απαντήσει ο κύριος Διοικητής. Όσον αφορά τον ενίο συντελεστή φορολόγησης, Έχουμε αυτό τον ενίο συντελεστή των προσωπικών εισοδημάτων, των φυσικών προσώπων εδώ και πολλά χρόνια. Έχουν γίνει πολλές πολιτικές συζητήσεις για το κατά πόσο πρέπει να τον αλλάξουμε. Ταυτόχρονα ένα από τα ζητήματα που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει είναι ότι ο φόρος των εργατικών στα εργατικά είναι λίγο υψηλότερος από ό,τι θα θέλαμε στο μέλλον θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια μεταβολή προς ε, φορολόγηση κατά κατηγορίες. Φυσικά έχουμε ήδη τέτοιες κατηγορίες γιατί υπάρχει αφορολόγητο εισόδημα για όλους τους ε, εργαζομένους. Αλλά θα μπορούσαμε να εισάγουμε ένα πιο προοδευτικό σύστημα διαφόρων κατηγοριών, όχι αυξάνοντας ε, το φορολογικό συντελεστή στα υψηλά εισοδήματα, αλλά μειώνοντας το φορολογικό συντελεστή για τα χαμηλά εισοδήματα προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός ε, φέτος. Αυξήσαμε το όριο του αφορολόγητου εισοδήματο που στη Λιθουανία εξαρτάται από το εισόδημά σας. Υπάρχει κάποιο τύπος, δεν είναι κάποιο σταθερό ποσό, πάγιο. Και αυτό επιτρέπει σε ανθρώπους που κερδίζουν ε, ε, πάνω από το 1,5% του μέσου μισθού να μην υποφελούνται από αυτό το φορολογητό. Έχουμε δηλαδή ένα, προοδευτικό, ένα σύστημα σε κατακατηγορίες αλλά χωρίς κατηγορίες συντελεστών φορολόγησης. Αυτή λοιπόν η κατηγοριοποίηση των φορολογητών εισοδημάτων ίσως να είναι μια μεθόδος που θα πρέπει να υιοθετήσουμε. Το μελετάμε. Τώρα όσον αφορά την διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, ε, αφενός εγώ θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί αυτή η διακυβέρνηση και να καταστεί πιο αποτελεσματική. Αφετέρου, βλέπω τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικότερα με το 6 και το 2-pack, δηλαδή τη σχετική νομοθεσία, με προληπτικό έλεγχο ε, των σχεδίων των κρατικών προπολογισμών. Είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση αυτά. Ορισμένες φορές στο Σουβουλέ Κοφίν ε, παρατηρούμε ότι κάποια συστήματα γίνονται τόσο περίπλοκα που χανόμαστε στο εσωτερικό τους. Κάπως λοιπόν πρέπει να διευθετήσουμε με πολύ έξυπνο τρόπο τις διαδικασίες αυτές ώστε χρονικά να συμπίπτουν για παράδειγμα. Θεωρώ ότι έτσι θα οδηγηθούμε σε καλύτερη διακυβέρνηση, πραγματικά. Αλλά μέχρι να υλοποιηθούν όλα αυτά θα χρειαστούν ακόμη 2-3 χρόνια θα έλεγα. Σε 2-3 χρόνια θα μπορέσουμε να έχουμε επιτύχει ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα δημοσιονομικού έλεγχου στην Ευρωζώνη. Παράλληλα διερευνάμε νέες ιδέες, νέες δυνατότητες βελτίωσης αυτής της διακυβέρνησης. Αλλά αυτή είναι η μόνη η δυνατή οδός κατά την άποψή μου. Τώρα όσον αφορά την αμοιβοποίηση των ε, χρεών Η κατάσταση στην Ευρωζώνη του 2007 ήταν αρκετά διαφορετική όταν η Λιθουανία έχασε το στόχο αυτό. Αλλά μπήκαν κάποιες χώρες ε, και έλαβαν ε, μια τεράστια όθηση φθηνού χρήματος που όπως αποδείχτηκε δεν ήταν ιδιαίτερα υγιές για τις οικονομίες τους. Αυτό είναι λοιπόν άλλο ένα κίνδυνο που διακρίνουμε εμεί για τη Λιθουανία. Ότι μπορεί να μεθύσει με φθηνά πιστώσει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί. Επιφυλακτικοί πριν χρησιμοποιήσουμε ε, πιστώσεις, ε, δανεικά δηλαδή. Έχουμε μάθει από παλιές υποθέσεις, ε, έχουμε αποκομίσει τα διδάγματα και είμαστε έτοιμοι να συμπεριφερθούμε πιο, ε, ε, να συμπεριφερθούμε πιο όρημα και υπεύθυνα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, λέει ο κύριος Βασίλειά Η πρώτη σα ερώτηση συνδέεται περισσότερο με τον τρόπο χρηματοδότησης των θηγατρικών των Σουηδικών τραπεζών στη Λιθουανία. Πρέπει να σας πω τώρα ότι μετά την κρίση του 2009 στη Λιθουανία έπεσε ραγδαία το ΑΕΠ. Και αυτό το μοντέλο χρηματοδότησης των σουηδικών ε, ε, θυγατρικών των τραπεζών στη Λιθουανία άλλαξε. Και μάλιστα με πολύ δραματικό τρόπο. Προηγουμένως, οι χορηγήσεις και τα δάνεια ερχόντουσαν κυρίως από τις μητρικές συστηγατρικές τράπεζες. Τώρα έχει αλλάξει το μοντέλο όπως είπαμε και τι σημαίνει αυτό. Ότι οι θηγατρικές εξαρτώνται περισσότερο από τις εγχώριες καταθέσεις. Άρα ο, ο, ο βασικός τρόπος και η κύρια πηγή ε, άντλησης ε, χαρτοφυλακίων ε, ε, χορηγήσεων και δανεισμού ε, είναι η μεδαπή αγορά, οι καταθέσεις των Λιθωνών. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει ε, στη διάρθρωση των τραπεζών μας. Αν το συγκρίνετε με την κατάσταση πριν την κρίση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μάλετιτς. Ε, ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό και τον Διοικητή και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για το κείμενο του στο μηνιαίο έντυπο του γραφείου μου, όπου μοιράστηκε μαζί μας τις εμπειρίες του. Μοιράστηκε με το κοινό στην Κροατία ε, τις εμπειρίες του να σας επενέσω για όλες τις πρόοδους που έχετε σημειώσει στα δημοσιονομικά και τις οικονομικές πολιτικές, ε, καθώς και στην εφαρμογή διαρθρωτικών ε, μεταρρυθμίσεων που στόχο έχουν να ενισχύσουν την αγορά εργασίας. Χάρη σε αυτές τις πολιτικές, από το 2011 και μετά ε, έχετε διαπιστώσει ανάπτυξη και είμαι βέβαιη ότι θα έχετε επιτυχία στην προσχώρηση στην ε, Νομισματική Ένωση το 2015. Ήρθατε σήμερα εδώ με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ε, και νομίζω ότι αλληλοσυμπληρώνεστε πολύ καλά ε, όσον αφορά τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που σας θέτουμε. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την συνεργασία σε θεσμικό επίπεδο ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα όταν μιλάμε για την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική συνεργασία αυτή είναι θεσμοθετημένη και πώς λειτουργεί όσον αφορά το πρόγραμμα. Επίσης, έχετε κοινά μέτρα για την χρηματοδοτική υποστήριξη επιχειρηματιών. Έχετε συνεργαστεί στην, ε, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή αυτών των μέτρων. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πράγματι ήταν χαρά μου να σας ε, δώσω το κείμενο. Ε, εργαστήκαμε μεγάλη προσοχή πάνω στο κείμενο αυτό. Χαίρομαι που έγινε τόσο θετικά αποδεκτό από εσά. Όσον αφορά τη συνεργασία, δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει επίσημη ε, θεσμική συνεργασία ανάμεσα στην κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα. Φυσικά έχουμε μία επιτροπή για την προσχώρηση στο ευρώ, κάτι που αποτελεί μάλλον εξαίρεση, στην οποία συμμετέχουν ο Πρωθυπουργό, ο Υπουργό Οικονομικών και ο Διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα. Ε, ανεπίσημα έχουμε πολύ καλή συνεργασία, ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα τη εισαγωγή του ευρώ. Όσον αφορά τα μέτρα υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτό είναι θέμα οικονομική πολιτική. Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας ε, δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα. Το θέμα αυτό αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της κυβέρνησης ως εκτελεστική ε, εξουσία, αλλά και του νομοθέτη, δηλαδή του Κοινοβουλίου. Πιστεύω λοιπόν ότι εμείς θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας ε, και η Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας έχει δική της εντολή. Αυστηρή εντολή Ίσως μπορεί ο διοικητής της τράπεζας να σας πει λίγα λόγια για αυτήν. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά τη συνεργασία σε θεσμικό επίπεδο ανάμεσα στον ε, Υπουργό Οικονομικών και την Τράπεζα της Λιθουανίας, φυσικά η Τράπεζα της Λιθουανίας έχει ειδικό νομικό καθεστώς. Είμαστε ανεξάρτητοι από την κυβέρνηση Ε, συμμετέχουμε στο δίκτυο κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν ειδικό καθεστώς. Στην περίπτωση της Λιθουανίας όμως, η κεντρική τράπεζα είναι ρυθμιστής και επόπτης του ε, χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στον τομέα αυτών ε, συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Οικονομικών. Όσον αφορά την νομισματική πολιτική, όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή έχουμε το ε, Συμβούλιο Συναλλάγματος από το 1994 και μετά, το οποίο σημαίνει ότι η Λιθουανία είναι χώρα εισαγωγών και έτσι λοιπόν ε, δεν ε, έχουμε πολλές επαφές στο θέμα αυτό με το Υπουργείο Οικονομικών. Όσον αφορά άλλα ζητήματα, όπως ανέφερε ο Υπουργό. συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά δημοσιονομικά θέματα ιδιαίτερα όσον αφορά ε, έναν ε, νέο νόμο που στηρίζεται στην ε, δεσμήτα 2 μέτρων και δεσμήτα 6 μέτρων που θα τεθούν σε ισχύ μάλλον από τις αρχές του επόμενου έτους. Τον ρόλο μας ως κεντρική τράπεζα, τον... πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας ως κεντρική τράπεζα είναι πολύ σαφής στο πλαίσιο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Σίμων, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε Υπουργέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω εδώ και επίσης να επαναλάβω αυτό που επανειλημμένως τόνισαν και οι συνάδελφοι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που καταφέρατε ε, να τα βγάλετε πέρα σε αυτό τον ανώμαλο δρόμο και το σκληρό για την ένταξή σας στην Ευρωζώνη την 1η Πρώτου 2015. Εποτείω ένα φόρο τιμής ε, στις θυσίες που κάνατε και τις προσπάθειες να ξεπεράσετε την κρίση τα τελευταία χρόνια. Τα είπατε και σήμερα. Κάτι που μου προκαλεί κάποιους προβληματισμούς το είπαν και οι συνάδελφοι, είναι κάτι που διάβασα ε, για, τον πληθυσμό και πώς αποδέχεται το ευρώ και βλέπουμε ότι η πλειονότητα ε, των Λιθουανών είναι κατά της ένταξης του ευρώ. Και αυτό μου έκανε εντύπωση, διότι τα τελευταία χρόνια κάνατε μεταρρυθμίσεις με πολύ μεγάλες θυσίες και προσπάθειες και θα θεωρούσε κανείς ότι, πώς να το πω, θα θεωρούσε ο λαό έτσι λιγότερο κακό σε σχέση με αυτά που έχει πάθει όλα αυτά τα χρόνια την ένταξή του στο ευρώ που αν, ε, ε, ενδεχομένω προκύψουν κάποιες ακρίβειε ή κάποια προβλήματα. Είπατε ότι θέλετε να ελέγξετε την άνοδο των τιμών, δεν θέλετε άμεση παρέμβαση και ταυτόχρονα θα κάνετε μια εκστρατεία έτσι υπέρ του ευρώ για την ενημέρωση τη κοινή γνώμη. Εγώ όμω θέλω να ρωτήσω κάτι παραπάνω. Παρά όλα αυτά που κάνει, ε, η πολιτική, ο κόσμος στην τσέπη του νιώθει και στο περιβάλλον του αν είναι κάτι για τον ίδιο καλό ή κακό. Εσείς πολύ συγκεκριμένα και βράχει πρόθεσμα, όχι μακροπρόθεσμα, τώρα, αύριο, τι περιμένετε από θετικές αλλαγές να γίνουν με την ένταξη ε, στο ευρώ, που να τη ζει ο κόσμος στο πετσί του για να αλλάξει ενδεχομένως και να γίνει πιο θετική η θεώρηση του κόσμου. Μια δεύτερη ερώτηση. Ε, χάρηκα που θέλετε να συμμετέχει περισσότερο το Κοινοβούλιο στην Τραπεζική Ένωση και στο νέο μηχανισμό εξυγίανση των τραπεζών. Ξέρετε στο παρελθόν πόσο ε, οξία ήταν η κριτική του Κοινοβουλίου για τις μεθόδους και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε ή θα δημιουργηθεί αυτό το ε, Ταμείο Εξυγείας Τραπεζών, ότι παραμένει διακυβερνητική μέθοδος. Και θα με ενδιαφέρε παρόλα αυτά να ακούσω τη γνώμη σας. Εάν στο μέλλον αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, πώς σκέφτεστε να καλλιεργήσετε τη σχέση σας με το Κοινοβούλιο και στο μηχανισμό διάσωσης και στο μηχανισμό σταθεροποίησης ε, και στο σύμφωνο σταθερότητας. Γενικά ε, έχουμε βρει ένα τρόπο συνεργασίας που δεν βοηθάει πάρα πολύ για το μέλλον της Ευρώπης αυτό το διακυβερνητικό σχήμα. Εσείς πώς προτίθεστε να βοηθήσετε ως μέλο τη Ευρωζώνης για να μετεξελιχθεί αυτή η κατάσταση ως αρμόδιος υπουργό. Θεωρείτε ότι τέτοια πράγματα μπορούν να επαναληφθούν στο μέλλον ή μήπως χρειαστεί και εσείς προτιμάτε έναν άλλον δρόμο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ναι, σύνθετες ερωτήσεις που κάνετε και περίπλοκες. Φυσικά η μηπω χρειαστει και εσεις προτιματε εναν ενός άλλου φυσικα η εισαγωγη ενος θα μπορούσε να έχει κάποιες ε, περιορισμένες βραχυπρόθεσμες συνέπειες, αλλά περιορισμένες μόνο. Όταν μιλάμε για τις θετικές ε, επιπτώσεις ε, για τη Λιθουανία θα είναι βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Ήδη από τώρα οι επενδυτές θεωρούν ότι είμαστε χώρα της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου του 2015 χωρίς ακόμα επίσημη απόφαση. Η υιοθέτηση αυτής της πρότασης από όλους τους υπουργούς του ΕΚΟΦΗΝ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εσάς ε, ή από τους επόμενους ε, από το επόμενο νέο κοινοβούλιο, τον Ιούλιο Αλλά αυτή η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος θα πρέπει να αποφέρει ωφέλη για όλους μακροπρόθεσμα. Φυσικά έχουμε τις ε, βραχυπρόθεσμες ε, οικονομίες ε, διότι δεν θα πληρώνουμε πλέον τέλη συναλλάγματο, χαμηλότερα επιτόκια, χαμηλότερου στόκους με την απομάκρυνση του κινδύνου υποτίμησης ε, όταν υπολογίζει κανείς την απόδοση μιας επένδυσης. Αυτά θα γίνουν άμεσα. Ε, εντός 7 χρόνων η Λιθωνική Τράπεζα έχει υπολογίσει ότι αυτό θα μπορούσε να αποφέρει 2 ε, δισεκατομμύρια λίτας, δηλαδή 700 εκατομμύρια ευρώ άμεσων ωφελών μετά από την εισαγωγή αυτή του ευρώ. Μείον φυσικά, γιατί να μην ξεχνάμε ότι έχουμε ωφέλη, αλλά από αυτά πρέπει να αφαιρέσουμε κάποιες δαπάνες που θα έχουμε αναγκαία. Για παράδειγμα για τη βελτίωση των συστηματών πληροφορικής και τα παρεμφέρει. Θα υπάρξουν λοιπόν ωφέλη. Πώς θα φανούν στο λαό μας δεν ξέρω. κάποιες βραχυπρόθεσμες ε, επιπτώσεις θα είναι φθηνότερες πιστώσεις ε, για δάνεια που έχουν ληφθεί στο τοπικό νόμισμα με προσαρμογή του επιτοκίου σε έναν εσωτερικό δίκτυ, σε έναν χώριο δίκτυ. Και... Επαναπροσαρμογή στο Euribor. Αλλά φυσικά Έχουμε δει τι έχει γίνει στους γείτονες και τις άλλες ε, χώρες Ευρωζώνης. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τα κυριοφέλη θα εμφανιστούν μακροπρόθεσμα. Φυσικά κάπως θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ώστε να πείσουμε την πλειοψηφία να υποστηρίξει το ευρώ. Όπως συνέβη στην Εστονία. Σήμερα το 78% του λαού της Εστονίας ε, είναι υπέρ του ευρώ. Ε, θα ήθελα να διορθώσω εδώ αυτό που είπατε. Αυτή η πλειοψηφία δεν είναι κατά. Είναι απλά επικριτική και επιφυλακτική. Δεν είναι υπέρ κατά της διατήρησης του σημερινού νομίσματος. Αυτό που θέλουν είναι να βελτιώσουν τις ζωές τους και εξακολουθούν να μην πιστεύουν ότι το ευρώ θα βοηθήσει σε κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να τους πείσουμε. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση για την SRM, την διακυβερνητική ε, συμφωνία. Ο ενιαίος ε, ε, μηχανισμός εξυγίανσης στο SRM, ο SRM δεν είναι, είναι περιορισμένου εύρους μέχρι να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί όλος ο μηχανισμός σωστά. Αποτελεί το αντικείμενο τριμερούς διαλόγου μεταξύ Συμβουλίου, ε, Επιτροπής και Κοινοβουλίου και για μένα Πρέπει σε όλες αυτές τις συζητήσεις, στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγένσης, όλες αυτές τις συζητήσεις να συνδεθούν με τις συζητήσεις ε, ε, ε, εκπόνησης μιας διακυβερνητικής συμφωνίας. Το Κοινοβούλιο βρίσκεται εκεί και συμμετέχει στην όλη διαδικασία. Ευχαριστώ κύριος Κλίντς. Ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά την πρώτη μου επίσκεψη στη Λιθουανία το 2006 όταν είχα την ευκαιρία να συζητήσω με καθηγητές και φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Βίλνιους για την εισαγωγή του ευρώ, που τότε, τότε θεωρείτο επικείμενη το 6. Δεν έγινε αυτό, διότι τότε παρόλο που πληρούσαν τα κλητήρια, ο πληθωρισμός ε, αναμενόταν ε, υψηλός και τελικά ε, αυτό επιδείχθη αληθές και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις τιμές ενέργειας. Και η κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια σήμερα. Ε, έχετε πολύ μεγάλη εξάρτηση από την ενέργεια, ιδιαίτερα από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης ε, πρόκειται να αποφασίσουν την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, οπότε δεν γνωρίζουμε αν η Ρωσία αποφασίσει να προβεί σε αντίπεινα και αν συμβεί κάτι τέτοιο μπορεί να αντιμετωπίσετε και πάλι κίνδυνο και σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι αφορά την ίδια τη διάθεση ε, και ενέργειας και τιμών. ερώτηση λοιπόν, έχετε σχέδιο Β για το πρόβλημα αυτό το ενεργειακό, αν προκύψει τίποτα, έτσι ώστε να μην διακυβευτεί η ένταξή σας στην Ευρωζώνη από τις τελευταίες εξελίξεις. Ένα δεύτερο που θέλω να ρωτήσω έχει να κάνει με μισούς και συντάξεις στο δημόσιο τομέα. Είπατε ότι πρόκειται να εντάξετε κάποιο είδους προοδευτική φορολόγηση την επόμενη, τα επόμενα δύο-τρία χρόνια. Είχατε όμως αρχικά σχεδιάσει να μειώσετε τους μισθούς και τις συντάξεις. Και εξ όσων γνωρίζω, το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο είπε αποκλείεται. Αυτό είναι αντισυνταγματικό ή παράνομο, δεν θυμάμαι τι είπε. Δεν επιτρέπεται να το κάνετε. Λοιπόν, και πάλι έχω την εξή ερώτηση. Τα επιπλέον έσοδα που ελπίζετε να αποκομίσετε με αλλαγή του φορολογικού συστήματος, με μια προοδευτική ε, ε, φορολόγηση, τελικά θα προκύψουν έτσι τα έσοδα ε, που είχατε προγραμματίσει ε, όταν ε, στην αρχή αποφασίσατε αυτά τα μέτρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Βόλφ. Όχι μόνο έχουμε ένα λαπτικό σχέδιο, αλλά μάλιστα το εφαρμόζουμε πολύ εντατικά. Σκοπεύαμε λοιπόν να έχουμε έναν σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το τέλος ε, αυτού του έτους. Ε, εργαζόμαστε όμως ε, πάνω σε επιπλέον συνδέσεις με την Πολωνία και με την Σουηδία στον ενεργειακό τομέα. Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα δηλαδή και στόχο έχουμε να αποφύγουμε την πλήρη εξάρτηση από μία πηγή ενέργειας που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι η ΚΑΣΠΡΟΜ. Θέλω όμως να αποφύγουμε και την εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τη Ρωσία. Πιστεύω λοιπόν ότι βράχει πρόθεσμα θα μπορέσουμε να ε, είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αυτό από μόνο του παίζει σημαντικό πολιτικό ρόλο ε, στις διαπραγματεύσεις μας με την ε, Gazprom και τους προμηθευτές μας από την Ανατολή. Έχουμε λοιπόν μία στρατηγική, η οποία αναφέρεται και στην έκθεση του Βέρνερ. Πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει. Όσον αφορά το αποτέλεσμα της ε, εσωτερικής αξιολόγησης που συζητήθηκε της υποτίμησης ε, και όσον αφορά τις ε, συντάξεις. Είχαμε απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου ότι δεν μπορούν να μειωθούν χωρίς ε, κατάλληλη αποζημίωση στο μέλλον και είχαμε περαιτέρω αποφάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου πριν από μία-δύο εβδομάδες Οι αποφάσεις έλεγαν ότι η ανάγκη για αποζημιώσεις θα πρέπει να συνάδει με την ικανότητα του δημοσίου τομέα να πληρώσει τέτοιες αποζημιώσεις. Νομίζω ότι αυτά είναι καλά νέα για μας. Μπορούμε έτσι να λύσουμε αυτά τα εκρεμή ζητήματα με σωστό τρόπο. Και έτσι σκοπεύουμε να προχωρήσουμε. Θα δούμε τι δυνατότητες θα υπάρξουν ε, στο μέλλον ε, για να λυθούν ε, αυτά τα θέματα αποζημιώσεων και θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Εάν βέβαια είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν τέτοια μέτρα στο μέλλον, θα το σκεφτούν αυτό οι μελλοντικέ κυβερνήσει, αλλά νομίζω ότι μιλάμε για ε, αρκετά μακρινό μέλλον. Κάποιοι οικονομολόγοι ίσως ε, να διαφωνήσουν μαζί μου, αλλά πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχουμε συγκεντρώσει κάποιες εμπειρίες σχετικά με το τι θεωρείται νόμιμο και τι όχι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι περικοπών των μισθών και μερικοί είναι νόμιμοι, συνάδουν με το Σύνταγμα, μερικοί όχι. Αυτές οι περικοπές ε, σύντομα με το σταγματικό δικαστήριο ήταν ε, παράνομες, ε, αλλά μπορούν να γίνουν αναλογικές μειώσεις στη Λιθουανία. Αυτά λοιπόν είναι καλά νέα για μας και θα... Είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίγκολτ έχει ζητήσει το λόγο. Αν δεν θέλει κανένας άλλος, θα τελειώσουμε. Ο κύριος Γκίγκολτ όμως. Ναι. Ευχαριστώ και εγώ να σας καλωσορίσω και να σας συγχαρώ. Ωραίες αποφάσεις παίρνετε και ωραία τα νέα που ακούμε. Ευχάριστα για όλα τα μέλη της Ευρωζώνης. Το μήνυμα ότι αυξάνεται ακόμα η Ευρωζώνη, μεγαλώνει. Είναι και πολιτικό το μήνυμα καθόλου ευκαταφρόνητο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν κάποιες ε, ανησυχίες που τις θεωρώ αρκετά υπερβολικές, διότι είστε ήδη στο δεύτερο μηχανισμό ισοτιμιών, ουσιαστικά είστε ήδη μέλος του ευρώ. Αυτό που κερδίζετε είναι η δυνατότητα να συναποφασίζετε για τη μοίρα σας. Δεν χάνετε τίποτα και όλη αυτή η φασαρία που γίνεται ε, είναι μάλλον συμβολική και υπερβολική. Γι' αυτό και πιστεύω ότι τελικά θα αλλάξει και ο κόσμος άποψη. Αν είχατε ρωτήσει τους Γερμανούς αν ήταν υπέρ του ευρώ και εκεί η πλειοψηφία κατά ήτανε. Στο μεταξύ είναι υπέρ βέβαια η πλειοψηφία των Γερμανών και έχουν καταλαγιάσει κάπως τα πράγματα, έχουν ησυχάσει. Σας ευχαριστώ. Μια σύντομη ερώτηση έχω. Είπατε ότι θα μπείτε και στην κοινή εποπτεία των τραπεζών, ε, είπατε ότι το είχατε και πρόθεση άλλωστε, και το δημοσιονομικό σύμφωνο αυτό τώρα το υιοθετείτε. Τι γίνεται με το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Τα περισσότερα κράτη της Ευρωζώνης συνεργάζονται και θα χαιρόμουν πάρα πολύ εάν ε, εκφράζετε την επιθυμία προσέγγισης αυτής της ενισχυμένης συνεργασίας και πώς το βλέπετε αυτό στην πορεία σας προς την Ευρωζώνη. Θέλετε να ενταχθείτε σε αυτό το μηχανισμό. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Φυσικά Καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε ήδη εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρωζάνη από το 2002 και έχουμε στη διάθεσή μας βέλτιστες πρακτικές για το πώς να συμπεριφερόμαστε σε δύσκολους καιρούς και μπορούμε να αναγνωρίσουμε και τους κινδύνους, ε, τις καλές εποχές. Ήταν πολύ καλό μάθημα αυτό για μας και ελπίζω να το μάθαμε σωστά. Τώρα όσον αφορά το το των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, δεν ε, έχουμε ακόμα αλλάξει την ε, επίσημη θέση. Δεν έχουμε υποβάλει επίσημα αίτηση για συμμετοχή. Στους επόμενους μήνες πιστεύω το ζήτημα αυτό το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα συζητηθεί σε κάποιες συναντήσεις του ΕΚΟΦΗΝ. Το πήρε το μαθήμα στην ατζέντα της Ελληνικής Προεδρίας. Νομίζω το Μάιο κάπου. Θα δούμε λοιπόν ε, τι πρόοδος έχει επιτευχθεί για τα ζητήματα αυτά. Από όσο εγώ γνωρίζω, είναι πολύ αργή η πρόοδος. Πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να δούμε, να σκεφτούμε πώς θα προχωρήσουμε, αλλά δεν υπάρχει ακόμα επίσημη απόφαση της λιθωνικής κυβέρνησης. Ευχαριστώ κύριε Δίκτα της Κεντρικής Τρέψης, θα να προσθέσετε κάτι. Όχι, δίνω τέλος το λόγο στον κύριο Λάνιεν. Μια σύντομη ερώτηση ε, που ε, μου ήρθε όταν μίλησε ο κύριος Γκίγκολτ που είπε ότι θα μπορείτε να συναποφασίσετε. Ε, θα είστε το 19ο μέλος και ε, ε, μειώνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, στη Γερμανία γίνεται λόγος, το θεωρώ σωστό, δεν θα το αναφέρω στην έκθεσή μου, αλλά σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών έχουν γίνει συζητήσεις και μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των μελών. έχουν τέσσερις μόνο με δικαίωμα ψήφου οι μεγάλες χώρες και οι μικρές ακόμα λιγότερους. Ε, πώς θα αλλάξει ο ρυθμός, κάθε μήνα θα είναι κάποιος άλλος, πώς το έχετε ρυθμίσει εκεί για τη στάθμιση των ψήφων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ορίστε. Θα σας δώσω πρώτα το λόγο αν θέλετε να συνοψίσετε. Όχι, ωραία, ο κύριος Διοικητής. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ καλή η ερώτησή σας και η απάντησή μου θα είναι σύντομη. Πιστεύω ε, θα έλεγα ότι οι διοικητέ, ακόμα και αν δεν έχουν ε, δικαίωμα ψήφου, ε, μπορούν να μιλήσουν. Έχουν φωνή και πιστεύω ότι μπορούμε να αναμένουμε η απόφαση για την προσχώρηση της Λιθουανίας ε, στη ζώνη του ευρώ να ληφθεί με βάση το, ε, το πρόγραμμα σύγκλησης. Από ό,τι γνωρίζω, οι περισσότερες αποφάσεις ε, λαμβάνονται με βάση τη συνένεση και ελπίζω αυτό να ισχύσει και σε αυτή την περίπτωση. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. 20 δευτερόλεπτα ίσως έχω στη διάθεσή μου. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Είσαστε οι εκπρόσωποι μας στην Ευρώπη. Η πολιτική σας υποστήριξη λοιπόν είναι πολύ σημαντική για μας. Και η προσωπική σας υποστήριξη αλλά και η πολιτική σας υποστήριξη για την προσχώρηση της Λιθουανίας ε, στην Ευρωζώνη θα περάσει πιστεύω και στο επόμενο κοινοβούλιο που θα πρέπει να ψηφίσει πάνω στο θέμα αυτό τον Ιούλιο. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της Ευρωζώνης βλέπουμε ένα κοινοβούλιο να συζητάει και το άλλο να αποφασίζει. Αλλά θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε όλα τα μέλη του νέου κοινοβουλίου να ψηφίσουν με καθαρή τη συνείδηση υπέρ της προσχώρησης στην Ευρωζώνη του 19ου αξιόπιστου εταίρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Βασίζομαι στην πολιτική σας υποστήριξη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Δικητά. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή λίγων δευτερολέπτων πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα για να ξεβγάλουμε τον Υπουργό και τον Δικητή. we move on. Mr. Langen, you are leaving? Werner. Κύριε Βέρνερ Λάγκερ, πού πάτε? Αν θέλετε να χαιρετήσετε εδώ τα στελέχη. We move on to next item of the agenda point 4, the preparation. Πάμε στο επόμενο θέμα, το 4. Είναι η έκθεση του κύριου Λάγκεν, πιθανή υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία εξέταση του σχεδίου έκθεσης, άτυπη είπαμε, Βέρνερ, έχει το λόγο. Οκ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Προεδρεύοντα, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Λιθουανίας και τον Υπουργό Οικονομικών για πολλά θέματα. Εδώ και λίγο καιρό ε, έχετε και την έκθεσή μου και μάλιστα μεταφρασμένη στις 3 Τρίτου υπευλήθη επίσημα. Τι λέω σε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Τα σημαντικότερα θέματα που συζητήσαμε και τώρα, βάσει των εκθέσεων μέχρι τώρα, είναι ε, ένα σαφές ναι, καταφατική απάντηση, αλλά έχουμε προβλήματα στοιχείων και προβλήματα ημερομιών. Τα στοιχεία τα τελευταία και τα πιο οριστικά θα τα έχουμε το Μάιο και προηγουμένως δεν μπορούμε να κάνουμε την οριστική αξιολόγηση. Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας και πριν τη συνεδρίαση είχαμε και διμερείς επαφές με τους δύο κυρίους που ακούσαμε μόλις και σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, τα οποία δεν είναι ακόμα επίσημα, η οικονομική κατάσταση θα εξακολουθήσει να σταθεροποιείται και δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, να αφισβητούμε γιατί η πρόγνωση του ε, χειμώνα να μην συνεχιστεί και την άνοιξη. Οπότε μάλλον πρόοδου θα κάνει προ το ευρώ παρά οπισθοδρόμηση η Λιθουανία στο επόμενο διάστημα. Ωστόσο, εμεί έχουμε ευρωεκλογέ τώρα. Γι' αυτό στην τελευταία συνεδρίασή μας που θα είναι μάλλον τον, 7 Απριλίου θα πρέπει να αποφασίσουμε και να ε, διαβιβάσουμε την απόφασή μας στο επόμενο κοινοβούλιο με το καλό αυτή είναι η αντικειμενική δυσκολία που έχουμε. Ε, τι σημαίνει αυτό μεταφρασμένο, ότι έχουμε σχετικά μικρή προθεσμία για ε, τροπολογίες. Η γραμματεία προτείνει τούτη εδώ τη βδομάδα. Έχω ακούσει όμως ότι υπάρχει μεγάλη ε, συνένεση και προθυμία των πολιτικών ομάδων να υπερψηφίσουν για να συνοδεύσουν τη Λιθουανία στην πορεία της προς το ευρώ. Επειδή όμως δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πραγματα αρων άρων-άρων και με τέτοιους ρυθμούς, γι' αυτό βάσει του σχεδίου έκθεσης να κάνουμε τροπολογίες προτείνω. Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών, θα το δούμε όταν έρθουν τροπολογίες και μπορούμε να τα ενσωματώσουμε όλα, αλλιώς αν χρειαστεί θα συνεδριάσουν και σκιώδεις. Και να ε, πω κάποια σύντομα πράγματα για την έκθεση αυτή η εισαγωγή ε, βασίζεται στα δεδομένα και τα στοιχεία σύμφωνα με τελευταία έκθεση σύγκλησης της 3ης Μαρτίου ε, ε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που ήταν ιδιαίτερα θετική. Είχαμε και άλλα θετικά στοιχεία για τη Λιθουανία, ακόμα και το Δούνου του δηλαδή τα λέει αυτά και συνηγορεί με την ένταξη της Λιθουανίας, καθόλου δεν την αμφισβητεί. Έχει χαμηλό πληθωρισμό η χώρα και μετά το 2009 που ξέσπασε η κρίση ε, κατέγραψε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μειώθηκε η ανεργία. Δεν υπάρχουν εντάσεις της εναλλαγματικής οτιμία με το ευρώ. Από το 2020 είναι ήδη συνδεδεμένη με το ευρώ ε, τα ονομαστικά επιτόκια είναι χαμηλά, τα κριτήρια του Μαστρίχτ πληρούνται, δεν υπάρχουν μακροοικονομικές ανισορροπίες που να διαπιστώνονται και η Βουλή της χώρας ήδη από το Γενάρη έχει προβεί σε αλλαγή της νομοθεσίας και επίκειται και μελλοντική αλλαγή. Τα είπε και ο διοικητής της τράπεζας ε, πώς θα γίνουν όλα αυτά και σε ό,τι αφορά την πρακτική εισαγωγή του ευρώ είναι όλα εγκαίρως στο χρονοδιάγραμμα. Σταμάτησαν και οι διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος του 2013. Υπάρχει το θέμα της υψηλούς, ε, ε, υψηλής συγγνώμη, εξάρτησης από την ε, ενέργεια και υπάρχει σχέδιο απαγκίστρωσης από την υπερβολική εξάρτηση και η ενεργειακή απόδοση. Στο σημείο 12 τα λέω αυτά και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν ήταν δύο τα πυρηνικά εργοστάσια Ιγναλίνα, αλλά ήταν ένα με δύο διαφορετικούς, τελείως ανεξάρτητους πυρηνικούς αντιδραστήρας. Πάνω από 1000 ΜΒ είναι μεγάλη αυτοί οι αντιδραστήρες που τροφοδοτούσαν τη Βαλτική. Ο πρώτος έκλεισε το 2006 και ο δεύτερος το 2009. Εγώ το 2008 την Άνοιξη πήγαμε την Επιτροπή Βιομηχανίας και με έπεισαν και θυμάμαι πάρα πολύ αυτά που είχε πει η κυρία Χάρμς τότε των Πρασίνων και θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τις συζητήσεις και τις ε, δεσμεύσεις του Ρώσου ε, διευθυντή εκεί που άρχισε σχεδόν να κλαίει. Έβαλε τα κλάματα γιατί είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε 300 εκατομμύρια για την ασφάλεια και ε, στο παρελθόν είχαμε περίπου 30 συμβάντα για κάθε αντιδραστήρα. Ε, τώρα έχουμε μόνο ένα και τώρα αυτό το, το παιδί μου το αγαπημένο που το έχτισα με τα ίδια μου τα χέρια και το μεγάλωσα τα τελευταία 30 χρόνια ε, και τώρα που λειτουργεί σωστά με αναγκάζουν να το κλείσω. Απλώς θα λέω αυτά γιατί στη Βαλτική ε, δεν ε, ήταν όλοι σύμφωνοι με τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα τμήμα της εξάρτησης από τη Ρωσία στα ενεργειακά θέματα έχει να κάνει ακριβώς με τον παροπλισμό της Ιγναλίνα. Το μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Ε, και θα το δούμε και αυτό είναι ε, μεγάλη μείωση της ενέργειας για όλη τη Βαλτική. Στο σημείο 15 έχουμε κάποια προσωρινά στοιχεία. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία βλέπουμε μείωση της ρευστότητας όπως ε, μας είπε σήμερα ο διοικητής ε, είναι σταθερή η κατάσταση και αντί για το 38,3% που αναφέρεται στο σχέδιο έκθεσής μου το ε, νεότερο νούμερο είναι 41,2%. Βλέπουμε λοιπόν, ε, έχουμε λοιπόν σταθερό ποσοστό εδώ και ακούσαμε διάφορες ε, ερωτήσεις. Ο κόσμος είναι κάπως επιφυλακτικός, αλλά όταν συνειδητοποιήσει ο κόσμος πόσο η προσχώρηση στο ευρώ θα ε, σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στην Ευρώπη και απέναντι ε, στη Ρωσία και στις σχέσεις της με τη Ρωσία. Πιστεύω ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αύξηση της αποδοχής ε, του κόσμου και όσον αφορά το τελευταίο σημείο και την Ρωσία, η Λιθουανία σε αντίθεση με την Εστονία και την Λετονία έχει μικρότερη ε, ρωσική μειονότητα και τους έχει δώσει λιθουανική υπηκότητα και έτσι η ε, ένταξη, η κοινωνική ένταξη ήταν μεγαλύτερη από ό,τι στα άλλα κράτη της Βαλτικής. Εγώ είμαι αρκετά βέβαιος ότι σε ένα χρόνο θα μπορέσουμε να δούμε την ε, προσχώρηση της Λιθουανίας στο ευρώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παδάρο, όχι. Άλτε, κύριε Στρεμόσα. Yes. Um, um, I hope. Ναι, ελπίζω και θέλω όλα, θα ήθελα όλα τα κράτη-μέλη να είχαν μπει στο ευρώ τόσο καθαρά όσο το πράττει η Λιθουανία. Ελπίζω λοιπόν ότι όλοι οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές θα υποστηρίξουν αυτή την εκθεσή και την ταχεία προσχώρηση της Λιθουανίας στην Ευρωζώνη. Κύριε Λάγγεν, θέλουμε να σας βοηθήσουμε στις εργασίες σας. Πιστεύουμε ότι όλα είναι εντάξει. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ομαλά μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ραμόν. Από τους πράσινους ο κύριος Πάσετ. Ευχαριστώ. Και εμείς ε, συμφωνούμε με την ανάλυση του κυρίου Σιγητή. Δηλαδή ότι η Λιθουανία βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να προσχωρήσει στην Ευρωζώνη. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Σιγητή για τον τρόπο με τον οποίο αποκρυπτογράφησε και εντόπισε και αναγνώρισε τις προσπάθειες της Λιθουανίας ε, για να συμμορφωθεί με τα κριτήρια σύγκλησης. Δεδομένων αυτών ε, πρέπει να πούμε και μια αλήθεια, ένα πρόβλημα που παραμένει, το οποίο γνωρίζετε μάλλον, Έχετε επιμείνει σε αυτό στην ομιλία σας. Ε, έχουμε μια εντύπωση ότι εμφανίζεται ένα νέο κριτήριο σύγκληση στην έκθεσή σας. Το πυρηνικό ζήτημα πρέπει να ξαναζητηθεί στη Λιθουανία ώστε να πληρεί τους όρους ε, για προσχώρηση στην Ευρωζώνη. Για μας το πυρηνικό θέμα, πέραν το ε, κατά πόσο πρέπει να συμπεριληφθεί όχι στο ενεργειακό μείγμα, δεν έχει θέση στις συζητήσεις περί προσχώρησης ε, στο νευροζώνη. Είναι εκτός θέματος, είναι άσχετο. Δεν συμφωνούμε να αποτελεί το πυρηνικό ζήτημα ένα ε, θέμα κλειδί στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προσχώρηση της Λιθουανίας στην Ευρωζώνη. Στο μεταξύ θεωρούμε ότι πράγματι θέτει το ενεργειακό ζήτημα στη Λιθουανία όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Υπάρχουν προσδοκίες εξέβρεσης λύσεων διασύνδεσης των ηλεκτρικών συστημάτων, ενεργειακή απόδοση, ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ναι, βέβαια, αλλά το να χρησιμοποιούμε αυτήν εδώ τη στιγμή την ευκαιρία της προσχώρησης της Λιθουανίας στο ευρώ για να επιμείνουμε ε, για επανεκκίνηση του προγράμματος ε, πυρηνικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μας φαίνεται ότι δεν έχει σχέση. Θα υποβάλουμε λοιπόν κάποιες τροπολογίες επί του θέματος ώστε η προσέγγιση του ενεργειακού ζητήματος να γίνει πιο ισορροπημένα. Παρομοίως θα θέλαμε η έκθεση να αναφέρεται στο ζήτημα της μετανάστευσης που πλήττει την ε, λιθουανική νεολαία. 500.000 Λιθουανοί, νέοι Λιθουανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους τα τελευταία χρόνια. Ναι λοιπόν ε, για την προσχώρηση της Λιθουανίας, αλλά όχι στο να προσθεθεί ένα επιπλέον κριτήριο η επανακίνηση της πυρηνικής ενέργειας στη Λιθουανία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέσετ, κύριε Σπάρα. Σας ευχαριστώ. Λίγα λόγια να πω. Εξήγησα τη θέση μου εξήγησα και τη θέση της ομάδας μου στις ερωτήσεις μου προς τον Υπουργό. Είμαστε υπέρ της έκθεσης αυτής. Ο Υπουργός παρουσίασε τη θέση της Λιθουανίας στον τομέα της ενέργειας. Καταβάλουμε προσπάθειες για την εισαγωγή αηφόρων πηγών ενέργειας, καταβάλουν προσπάθειες για τη δημιουργία ε, σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και ε, όσον αφορά την ε, κοινωνική ένταξη των Ρώσων, η Λιθουανία έχει λιγότερους Ρώσους από ότι η Εστονία και η Λετωνία. Ο κύριος ο, ο συνάδελφος από τους Πασίνους ε, δεν ε, με κατάλαβε καθόλου. Πουθενά δεν λέει ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί προπόθεση. Απλά ζήτησα κατανόηση διότι τα ενεργειακά θέματα δεν λύνονται τόσο ε, εύκολα λόγω του παροπλισμού δύο πυρηνικών μονάδων. Το πώ ε, η Λιθουανία και η Βαλτική γενικά θα λύσουν το ενεργειακό θέμα στο μέλλον ε, θα το αποφασίσουν μόνες τους ε, οι χώρες αυτές. Δεν αναφέρεται τίποτα στην εκθεσή αυτή, απλά είπα ότι η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο έχει αυξηθεί μετά τον παροπλισμό των πυρηνικών μονάδων και γι' αυτό θα πρέπει να επιδείξουμε ιδιαίτερη κατανόηση όσον αφαιρώ την ενεργειακή πολιτική των βαλτικών χωρών. Αυτή ήταν η παρατήρησή μου. Απλά ε, δεν ήθελα να ξεχαστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βοηθήσει στην ε, περίπτωση αυτή, στο θέμα το, της ενέργειας. Ε, και αυτό έχω αναφέρει στο σημείο 12. Η δεύτερη μου παρατήρηση όσον αφορά τους νέους. εξέτασα ε, το θέμα. Κοίταξα τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τις αρχές του 2014 και η Λιθουανία έχει το υψηλότερο ποσοστό ε, αποφύτησης ηλικίου στην Ευρώπη, 94,5% για τις γυναίκες και 92% για τους άντρες, το οποίο σημαίνει ότι το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί κίνητρο για τους ε, νέους ε, στην ε, δύσκολη οικονομική κατάσταση να μεταναστεύσουν σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2004. Και για τις χώρες της Βαλτικής ισχύει λοιπόν ότι θα υπάρξει επιστροφή όταν βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια προσωρινή κατάσταση αυτή, δεν πιστεύω ότι είναι μόνιμη, είμαι αισιόδοξο στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Βέρνερ. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 20 Μαρτίου. Η συζήτηση των τροπολογιών θα γίνει στις 7 Απριλίου, η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΚΟΝ στις 7 Απριλίου επίσης και για προφανείς λόγους η Ολομέλεια δεν ξέρουμε πότε θα ψηφίσει. Ωραία. Όπως όλοι γνωρίζετε, έχουμε οικονομικό διάλεκτο και ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μοσκοβισή που έχει αναβληθεί για τέταρτη φορά παρακαλώ. Και ε, ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Όχι δεν ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται αφού αναβλήθη. Θα το ξαναπούμε αύριο στις 9 το πρωί για να συζητήσουμε το θέμα της Κροατίας για την προσχώρησή της Σύμβασης Σύμβαση της 23 Ιουλίου 1990 κτλ. Για την εξάλληψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση ορθώσεως των κερδών σε επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο.